βίωσαν. Θα μπορούσαμε λοιπόν να συσχετίσουμε το γεγονός αυτό και να ε, αποτίσουμε φόρο τιμής και σε αυτούς τους αλίες. Ευχαριστώ. Βεβαίως, συνάδελφε, συμφωνούμε απολύτως ότι θα πρέπει να εκφράσουμε τη θλίψη μας και για την προκείμενη περίπτωση. Πρακτικά, λοιπόν. Κύριε Σίμψον, θέλετε να πείτε κάτι. Πρόεδρε, θα ήθελα να στείλετε ένα τεχνικό στο 176 γιατί το μηχάνημα που έχω μπροστά μου δεν λειτουργεί καθόλου. Άμεσα κύριε Σίμψον. Τα πρακτικά λοιπόν της συνεδριάσεως της, της Τετάρτης 18ης Ιανουαρίου έχουν εγκριθεί και μάλλον συγγνώμη σας έχουν κατανεμηθεί, υπάρχουν σχόλια, όχι άρα θεωρούνται εγκεκριμένα. η ε, δήλωση Κάντικ και ε, λοιπόν η υπαριθμών 0041 κάθετος 2011 έχει ε, πετύχει τις υπογραφέ των περισσότερων μελών και επομένω σύμφωνα με το άρθρο 123 του κανονισμού θα μεταδοθεί σε όλους και θα προωθηθεί και επομένω θεωρείται εγκεκριμένη ο κύριος Κάντεκ για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, αδιαφυσβήτητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα λάβει υπόψη της αυτή τη γραπτή δήλωση και έτσι ε, θα λάβει υπόψη της αυτό το πρόβλημα των ευρωπαϊκών ακτών. Οφείλουμε να καταρτήσουμε ένα ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης εναντίον της διάδοσης ε, και της εξάπλωσης όλων αυτών των φυκιών, τα οποία λειτουργούν παρασιτικά. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι με βοήθησαν εδώ στο Στρασβούργο αλλά και τις προηγούμενες εβδομάδες. Εδώ στο Στρασβούργο που αισθανόμαστε όλοι τόσο καλά, αγαπητοί συνάδελφοι. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Λένιτσακ από πλευρά Σοσιαλιστών Δημοκρατών, τον κύριο Τρεμόπουλο από πλευρά Πρασίνων και τον ε, κύριο Τζανόνι από πλευρά Φιλελευθέρων. Ευχαριστώ όλους σας, αγαπητοί συνάδελφοι. Συγχαρητήρια η γραπτή δήλωση 0037-2011 που έχουν υποβληθεί από τον κύριο Δανέλη και λοιπόν όσον αφορά το σύμφωνο των νήσων έχει δεχτεί τις ε, ε, υπογραφές της πλειοψηφίας των μελών.